Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, υπεύθυνη για τον ανταγωνισμό Επίτροπο κυρία Φεστάγκερ και να την ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησής μας εδώ θα συζητήσουμε ε, την ε, υλοποίηση των συστάσεων που έκανε το Κοινοβούλιο στη διάρκεια αυτής της θητείας. Which Είμαι σίγουρος ότι θα πείτε ότι δεν θα ε, ε, συζητήσετε για θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί. Αλλά βέβαια εσείς ξέρετε και ποια είναι τα σημαντικά θέματα για μας και ποια μας ενδιαφέρουν, οπότε θα σας ζητήσω να πάρετε το λόγο και να κάνετε μία δήλωση που δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά όμως. Well, first of all, thank Uh, uh, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο της Επιτροπής Τάξη. Ευχαριστώ δε ιδιαιτέρως ε, για την εμπλοκή σας, ε, για την οργάνωση της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης, γιατί νομίζω ότι αυτό αυτά τα ζητήματα ενδιαφέρουν τους πάντες, ενδιαφέρουν τους επιχειρηματίες, ενδιαφέρουν τους πολίτες, ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Διότι εάν κανείς δουλεύει σκληρά όπως οι Ευρωπαίοι πολίτες και πληρώνεις και τους φόρους σου, ε, οπωσδήποτε θέλεις ε, να βλέπεις τι γίνεται με τα χρήματα αυτά. Επίσης, εάν είσαι επιχειρηματίας, ε, θέλεις ε, ε, και πληρώνεις και τους φόρους σου, θέλεις να πληρώνουν και οι ανταγωνιστές σου και να συμβάλλουν και αυτοί στην κοινωνία. That, uh, uh, large, uh, companies Δεν μιλάμε μονάχα για μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ε, πόρους ε, που θα πρέπει είτε να μην πληρώνουν είτε, είτε μάλιστα και να έχουν ειδικό καθεστώς. Εδώ και τέσσερα χρόνια στην ε, ε, στην δημοκρατική μας διαδικασία έχουμε προωθήσει πολλά στοιχεία έτσι ώστε να γίνει απόλυτα δύσκολη η φοροαποφυγή. 14 μάλιστα ε, νομοθετήματα αφορούν ε, νέα στοιχεία τις ε, τελευταίες δύο δεκαετίες και βεβαίως κατά την έννοια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά του Κοινοβουλίου γιατί κρατάει ένα ρυθμό εντατικό και γιατί και οι πολίτες βλέπουν συγκεκριμένα έργα. Ευχαριστώ ε, και τους ε, βουλευτές ε, που έχουν που έχουν υποβάλει τέτοιες ψηφίσματα συγγνώμη, και γνωμοδοτήσεις. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει και η δουλειά μας θα πρέπει να συνεχιστεί. είναι η στιγμή να μην δείξουμε αυταρέσκεια, να μην ε, επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και τι χρειάζεται να κάνουμε για το μέλλον. Και η συνέχιση των εργασιών μας έχει να κάνει και με τις κρατικές βοήθειες και τη σχετική δουλειά μας. Την περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για την βελγική εξαίρεση για τον ε, επιπλέον φόρο για τις πολυεθνικές, τον ειδικό φόρο για τις πολυεθνικές. Καλύπτονται κάποιες πολυεθνικές που μπορούν μέχρι 90% να μειώσουν το φορολογήσιμο τζίρο τους. 90% το δικαστήριο ε, υποστήριξε πλήρως το ότι η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των φορολογικών μέτρων που θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κρατική βοήθεια. Και αυτό είναι σημαντικό διότι η, κατηγορία όσων ε, ήθελαν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ε, στην ε, ε, υπόθεση αυτή έλεγαν ότι η Επιτροπή δεν έχει καμία δουλειά. Όμως η οι εταιρείε δεν έχουν πρόβλημα όταν πληρώνουν του κανονικού του φόρου. Τότε δεν είναι φορολογήσιμε από άλλε. Όμω το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να έχουμε ε, αποφασίσει την βελγική εξαίρεση ω γενικό πρόγραμμα κρατική βοήθεια. Κατά την άποψη του δικαστηρίου, η δίκηση του δικαστηρίου είχε ένα δικαίωμα διακριτική αυχέρεια για να αποφασίσει υπό ποιε προποθέσει η εξαίρεση μπορεί να δοθεί στι πολυεθνικέ που την ζήτησαν. Βάσει της απόφασης, η διακριτική αυτή ευκαιρία σημαίνει ότι οι εξαιρέσεις δόθηκαν σε τρόπο ατομικό και όχι ε, γενικά και καλύπτοντας τους πάντες. Οπότε το δικαστήριο ενίσχυσε την απόφαση του δικαστή της Επιτροπής να θεωρήσει ότι η φορολογία είναι ένα γενικό σύστημα. Δεν εξέφρασε άποψη για το αν οι επιμέρους εταιρείε ενισχύονται από κρατική βοήθεια ή όχι. Πάντως το δικαστήριο συμφώνησε με την Επιτροπή ότι η βελγική εξαίρεση δεν φαίνεται να επιδιώκει το στόχο της αποφυγής της διπλής φορολογίας των σχετικών κερδών. Και αυτό με τη δικαιολογία ότι αυτό είχε χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το Βέλγιο για να δώσει τις προλογικές εξαιρέσεις. Οπότε βλέπετε ότι η απόφαση είναι κάπως ανάμεικτη στα συναισθήματά της και στα όσα προβλέπει. Θα πρέπει λοιπόν εμείς αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα. Η απόφαση εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη, οπότε έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο, αλλά βεβαίως θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια παγιωμένη αρχή. Εάν ε, η φορολογία για τις εταιρείε είναι επιλεκτική, είναι κρατική βοήθεια και είναι παράνομη. Επίσης, αυτή την αρχή την ακολουθούμε και στις υπόλοιπες 7 αποφάσεις μας, όπου αναλύσαμε επιμέρους αποφάσεις και τις μελετήσαμε και για αυτές ζητήσαμε την ανάκτηση περίπου 15 δις ευρώ σε που δεν είχαν καταβληθεί από εταιρείε. Θα θυμάστε ότι το μεγάλο όγκος αυτού ήταν ε, το θέμα της Apple. Μετά συνεχίσαμε τις σχετικές μας έρευνες και τον περασμένο μήνα ξεκινήσαμε μια έρευνα για την Nike στις κάτω χώρες και επικεντρωθήκαμε στη φορολογική μεταχείριση δύο ε, Ολλανδικών εταιριών που ε, έχουν 2.000 εργαζομένους και φαίνεται ότι προωθούν την μάρκα Nike σε όλη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ειδικέ ε, μεταχειρήσεις για την εταιρεία Nike, φαίνεται ότι αυτές οι εταιρείε έτυχαν τη μεταχείρισης εταιρεών που δεν έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στις κάτω χώρες. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή ανησυχεί ότι αυτές οι πληρωμές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα των εταιρεών αυτών ή την οικονομική πραγματικότητα. Εάν αποδειχθεί αυτό, ε, όλος ο όμιλος Nike μπόρεσε τεχνικά να μειώσει τους φόρους του για ένα μεγάλο μέρος των κερδών της στην Ευρώπη, των κερδών του μάλλον. Συνεχίζονται επίσης οι ε, εξετάσεις των υποθέσεων για την IKEA, την IKEA για την ελεύθερη ζώνη της Μαδέρας και για τις εταιρείε και τις ειδικέ ε, διευθετήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως δεν υπάρχει υπόθεση που να μην είναι προτεραιότητά μα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά του να καθορίσουν φορολογικές προτεραιότητε και να μην αποφύγουμε τη συζήτηση για τις κρατικές βοήθειες σε πρώτη φάση είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τους περιορισμούς για την επιβολή των κρατικών βοηθειών σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι περιπτώσεις κρατικής βοήθειας με εταιρείε που λαμβάνουν επιλεκτικά πλεονεκτήματα, ενώ άλλοι όχι, είναι ένα θέμα. Όμως μόνο με την καλύτερη φορολογία και τους σχετικούς κανόνες μπορούν να επιληθούν ε, μόνιμα κάποια προβλήματα και να κλείσουν τα κενά, να καλυφθούν τα κενά που όλοι εκμεταλλεύονται, τα παραθυράκια αυτά. Οι κανόνε για τι κρατικέ βοήθειε και οι σχετικοί κανονισμοί πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα για να γίνει δίκαιη η φορολογία. Βλέπουμε να επιτελείται πρόοδο. Για να ονομάσω μερικές περιπτώσεις... η Κύπρος και το Λουξεμβούργο άλλαξαν τους φορολογικού του κανόνε για τις χρηματοοικονομικές εταιρείε. Η Ιρλανδία κατήργησε το διπλό Ιρλανδικό φόρο, το σχετικό αυτό σύστημα. Οι κάτω χώρες ξεκίνησαν μια ευρεία φορολογική μεταρρύθμιση και μόλις εγκριθεί οι φορολογικές αρχές θα ε, λαμβάνουν φορολογικέ αποφάσει μόνο για πραγματικέ επιχειρηματικέ δραστηριοποιήσει και δραστηριότητε και όχι μόνο για, και όχι για εικονικέ εταιρείε. Και επίση δεν θα γίνονται αποδεκτέ ε, φορολογικέ συμφωνίε που θα εμπλέκονται φορολογική παράδειση. Επίση θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό ετησίω για την προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για τις φορολογικές συμφωνίες. Επίσης, συστηματικά αναθεωρούμε και κοιτάζουμε τις πρακτικές των φορολογικών συμφωνιών σε όλη την Ένωση. Και αυτή η προσπάθεια μας έδωσε κάποια καλά πορίσματα ως προς το πώς να θέσουμε φορολογικές προτεραιότητες σωστά. Η Γερμανία, λόγου χάρη, στις φορολογικές συμφωνίες και σε όσου έχουν πληγεί από τι διευθετήσει τη για τι πολυεθνικέ δίνει υποζημίωση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μια χώρα να δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάποιε εταιρείε που να πλήξουν αυτά τα φορολογικά εισοδήματα μια άλλη χώρα. Στην Αυστρία κάθε φορολογική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τι φορολογικέ αρχέ και το top management μια ε, ε, φορολογική αρχή πρωτού ε, εγκριθεί. Και ενώ σε πολλά κράτη-μέλη απλώς γίνεται το προφανές, ε, δηλαδή κοιτάζουν ε, τα στοιχεία πριν ε, εγκριθεί μια φορολογική συμφωνία, και κοιτάζουν απλώς τους αριθμούς περί του τζίρου που τους δίνουν οι εταιρείε. Δεν ασχολούνται με την οικονομική πραγματικότητα και το αν οι αριθμοί αυτοί ανταποκρίνονται σε πραγματικά στοιχεία. Ούτε χρησιμοποιούν πάντα εξωτερικού εμπειρογνώμονε. Με αυτέ τι αρχέ οι ε, φορολογικές συμφωνίες ή η πλειοψηφία τους ε, ουσιαστικά εκπληρώνουν το σκοπό τους για να υπάρχει ασφάλεια για τις εταιρείες για το φορολογικό τους χρέος. Και βεβαίως ε, βάσει και της οικονομικής πραγματικότητας και για να μην μπούμε στο πεδίο των παράνομων κρατικών βοηθειών. Αυτό είναι κάτι καλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κλείνει τώρα τέσσερα χρόνια πολύ σκληρής δουλειάς για την ε, δίκαιη φορολογία. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και την αφοσίωση που δείξαμε για να πετύχουμε αυτό το σκοπό, νομίζω καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα ρυθμό που ίσως είχε κάπως χαθεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Διότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Και ελπίζω ότι κι εσείς θα μας ακολουθήσετε και στην υλοποίηση. Θα δείξετε την ίδια αφοσίωση για την ε, υλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Διότι νομίζω το πλέον σημαντικό είναι να σεβαστούμε το νομοθέτη φροντίζοντα να υλοποιηθεί η νομοθεσία. Είναι δύσκολο να εγκρίνουμε νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στα θέματα τα φορολογικά, διότι απαιτείται η ομοφωνία. Όμω οι δυσκολίε δεν πάβουν μόλι ε, ληφθεί μια απόφαση. Η υλοποίηση και η εφαρμογή είναι ένα άλλο θέμα. Εκεί φαίνεται το κατά πόσον η νομοθεσία κόστησε πολλά και σε κόπο και σε προσπάθειες. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα ζητήσει να υπάρξει σωστή υλοποίηση τη νομοθεσία που εγκρίθηκε. 14 νομοθετήματα, σημαντικά θεωρώ εγώ, πρέπει να δούμε πώ υλοποιούνται. Αλλά στη φάση τη παρακολούθηση και τη ε, εφαρμογή του, στα κράτη-μέλη θα δοκιμαστούν το βασικό πλεονέκτημα της δουλειάς που έχουμε κάνει πάντως είναι ότι η φορολογική δικαιοσύνη δεν είναι πλέον ταμπού. Ο καθένας μπορεί να το συζητάει και ο κάθε πολίτης το προσδοκά. Είναι κάτι που το συζητάμε και γι' αυτό έχουμε αναλάβει δράση προκειμένου να το πετύχουμε. Και αυτό βεβαίως είναι και το πώς θα έπρεπε να έχουν τα πράγματα. και για τις επιτροπές σας, τις επιτροπές τάξε, έχουμε αυτό το νέο εργαλείο, έχουμε αυτήν την ανοιχτή προσέγγιση. Η φορολογική δικαιοσύνη έχει γίνει το επίκεντρο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Και επ' αυτού θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά έχουμε αυτόν τον απλό και πολύ λογικό στόχο όλοι να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους στους φόρους. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πέτροπα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι η νομοθεσία η οποία εγκρίνεται θα πρέπει να υλοποιείται, να εφαρμόζεται σωστά. Αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα και όπως είπατε τα 14 νομοθετήματα τα οποία εγκρίθηκαν την τελευταία πενταετία, πιο πολλά από την προηγούμενη 20 ετία συνολικά, είναι παρόμοια με αυτά που δικαιολόγησε και ο Επιτροπός Μοσκοβεσία από δική του πλευρά. Και αυτό σαφώς επιβεβαιώνει ότι η μάχη, ο αγώνας για τη δίκη φορολόγηση έχει πλέον Έχουμε τώρα πέντε λεπτά για ερωταπαντήσεις. Ερωτήσεις στον ενός λεπτό. Και μετά υπόλοιπο χρόνο. Ο κύριο Μάιερο, εισηγητή από πλευρά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Και ξέρετε πόσο εκτιμώ την εργασία σα και τη σαφήνεια του μηνύματο που στέλνετε. Αυτό είναι σαφέ. Έχω τρία ερωτήματα. Καταρχάς όμως θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω το εξή. Είναι σημαντικό να υπάρχει συμφωνία από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και από τις διάφορες χώρες στο θέμα αυτό της καταπολέμησης της ε, φοροαπάτης. Κατά δεύτερον, μάλλον πρώτη ερώτηση, κάνετε εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό, αλλά μήπως δεν θα πρέπει να κάνουν και άλλοι τη δουλειά τους ε, Μήπω και άλλοι δηλαδή έχουν υποχρέωση να κάνουν τη δουλειά τους και να μην την κάνετε εσεί γι' αυτό σε ό,τι αφορά τον κωδικά δοντολογία. Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν σωστε λύσεις, γιατί σε πολλε περιπτώσεις δεν αρκεί η δική σα προσπάθεια. Κατά δεύτερον, χαίρομαι που το Συμβούλιο κατάφερε να περάσει κάποια νομοθετήματα. Δυστυχώ, τα πιο σημαντικά νομοθετήματα όπως το και τα λοιπά, ε, για την ψηφιακή νομοθεσία. Αυτά είναι στο πάγο. Το CCBD πιστεύετε ότι θα προορίσει τον κίνδυνο των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ακόμα και αν σημειωθεί πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέμαι σε τι βαθμό λαμβάνουμε υπόψη και την παγκόσμια διάσταση, γιατί τίθεται θέμα ανταγωνισμού, το, οι προσπάθειες ε, για την άμεση φορολόγηση δεν είναι ευρωπαϊκά ζητήματα αυτά μόνο, είναι παγκόσμια ζητήματα. Σε τι βαθμό λοιπόν πιστεύετε ότι χρειάζεται παγκόσμια πρόοδος και ελπίζουμε ότι θα συνδράμει και ο ΑΣΑ προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Απάντηση. Το πρώτο σημείο που θέσατε είναι μια ερώτηση που Μάλλον είναι ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων από πολλέ διαφορετικέ ε, πολιτικέ σκοπιέ. Και αυτό θεωρώ καταδεικνύει με σαφήνεια πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και καταδεικνύει άλλωστε ότι η φορολογική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο ασπάζονται και περιμένουν από εμά όλοι οι πολίτε όλη τη Ένωση κατά πόσον οι άλλοι τώρα θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω πράγματα. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε πριν από κάποια χρόνια ήταν το εξή. Όταν κάναμε την πρόταση, η οποία πλέον εγκρίθηκε για την αυτόματη αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων σε θέματα αφορολογία, κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι υπάρχει ήδη νομοθεσία η οποία επιτάσσει συνεργασία. Ναι, αλλά δεν συνέβαινε αυτή η συνεργασία. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα από πλευρά μα ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ε, ταχύτητα που έχουμε συγκεντρώσει για να αλλάξει και η νοοτροπία. Γιατί είναι παράδοξο ότι ναι, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει το πλαίσιο για τη συνεργασία, αλλά δεν χρησιμοποιείται και πρέπει να γίνει ένα επιπλέον βήμα σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για να υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, των οποίων θα έπρεπε η ανταλλαγή να αποτελεί ένα φυσιολογικό και αυτόματο φαινόμενο. Είναι παράδοξο ότι σε κάποιες περιπτώσεις μας ε, κατηγορούν ότι υπερβάλλουμε σε ό,τι φορά την νομοθεσία. Αλλά τι άλλο να κάνουμε στην περίπτωση την προκειμένη, πέρα από το να δώσουμε ακόμα μία όθηση. Άρα με τη νέα αυτή νομοθεσία ελπίζουμε να υπάρξει μία νέα νοοτροπία για το πώ λειτουργούν οι φορολογικέ αρχέ στα διάφορα και το πώ συνεργάζονται. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία. Η συνεργασία, ξέρετε, αποτελεί και τη βάση των τριών προτάσεων τις οποίες συζητάτε. Ψηφιακή νομοθεσία, μια κοινή βάση φορολογίας και η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Αυτά που θίξατε τα θέματα. Αυτά, ξέρετε, θα απλοποιήσουν τον τρόπο λειτουργία των ε, έντιμων μικρομεσαίων εταιριών θα καταστήσουν πολύ πιο εύκολες τις περιπτώσεις διατησίας και θα διευκολύνουν την σύμβολη στην κοινωνία. Και συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικά τα τρία αυτά νομοθετήματα. Πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό στην Ευρώπη επαφίεται να κατανοήσει ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αυτή είναι ουσιαστικά η όθηση την οποία προσπαθούμε να δώσουμε τώρα. Ιδάλλως, ε, πέραν από την ψηφιοποίηση, ε, αυτά τα νομοθετήματα δεν θα ήταν τόσο σημαντικά όσο είναι. Ξέρετε ότι ο συνάδελφος Μοσκοβισή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα προκειμένου αυτά να επιτευχθούν στο τέλος της θητείας. Προφανώς υπάρχει η παγκόσμια διάσταση. Προφανώς και γι' αυτό συνεργόμαστε, συνεργαζόμαστε τόσο πολύ με τον ΩΣΑ. Και ο ΩΣΑ σημειώνει πρόοδος και στην ε, ψηφιακή νομοθεσία και είδαμε ότι κάποιες ε, από τις τελευταίες πρόσφατες ιδέες συνάδουν με τον τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό. Εξακολουθώ φυσικά να πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή όθηση εντό του ΑΣΑ προκειμένου να προωθηθούν κάποια ζητήματα, προκειμένου να πετύχουμε γρήγορα κάποιες λύσεις. Γιατί αν είναι κατακριματισμένη η Ευρώπη, πιστεύω, δεν θα υπάρχει τόσο η αίσθηση του κατεπήγοντος και στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του ΟΣΑ. Η άλλη πλευρά της φορολογικής δικαιοσύνης είναι οι επιδοτήσεις, κατά αυτόν επιδοτήσεις που μπορούν να έχουν ε, πολλές διαφορετικές μορφές, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταχείριση, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ε, υπάρχει στον ανταγωνισμό αν έχει την κυβέρνηση από πίσω που σε υποβοηθά, που σου δίνει επαρκή χρηματοδότηση και έρχεσαι τελικά να ανταγωνιστείς με εταιρείε εδώ, οι οποίες στέκονται μόνε του στα πόδια. Έτσι λοιπόν με την Κίνα γίνεται μια συζήτηση σε διαφορά τις επιδοτήσεις. Η Σεσίλια Μάλμστρομ συνομιλεί με τους Ιάπωνες και τους Αμερικανούς, με, τον Παγκόσμιο, με την παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου. Προσπαθούμε λοιπόν και εκεί να δείξουμε μια ηγεσία, γιατί προφανώς και υπάρχει αυτή η παγκόσμια διάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεπέ. Και σας παρακαλώ να τηρήσουμε το πεντάλεπτο, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές. Ο Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και την ε, Επίτροπο ε, Φεστάγκερ και για την δουλειά που έχει κάνει, αλλά ε, και γιατί ανέφερε τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Αναφερθήκατε και στα 14 νομοθετήματα. Αυτό που είναι σαφές και το είπατε και εσείς και είναι πολύ σημαντικό, είναι η υλοποίηση του θεματολογίου για την φορολογία. Θυμάμαι, ας πούμε, ε, στην έκθεση πάνω είχαμε ακριβώς αναφέρει αυτό το θέμα και ότι η υλοποίηση θα πρέπει να γίνει από την Κομισιόν γιατί και στα, στο ξέπλυμα βλέπουμε ότι η ικανότητα, μη, η μη ικανότητα μάλλον εφαρμογή είναι ε, από τους πιο σημαντικούς φόβους που έχουμε. Ελπίζουμε ότι και η επόμενη Κομισιόν, η επόμενη Επιτροπή θα προχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. αποτελεσματική λοιπόν υλοποίηση. Να σας ρωτήσω, ε, υπήρχε και το, η υπόθεση McDonald's του Λουξεμβούργου. Πόσο πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις, τα παραθυράκια που υπάρχουν. Γιατί στην περίπτωση του McDonald's του Λουξεμβούργου δεν ήταν ακριβώς παράνομο, ήταν ένα είδος αποφυγής διπλής ε, φορολόγησης. Αλλά ε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει ε, ένα ίδιο επίπεδο για όλους και ορθός ανταγωνισμός. Επίσης, ε, λέτε ότι μπορούν να δοθούν ε, εξαιρέσεις ε, για έρευνα και ανάπτυξη και όχι παροχές ή εκπτώσεις. Ναι, αλλά ξέρετε ότι μερικές φορές ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορεί κανείς να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την έρευνα θα πρέπει να δούμε το θέμα από πλευράς ανταγωνισμού, από τη σκοπιά μάλλον του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρξει και η ανάπτυξη και η έρευνα και η καινοτομία, χωρίς όμως ε, να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κανείς, να προστρέξει σε αυτό το ε, εργαλείο, το οποίο δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ο Πιέρ Μοσκοβισή μάλλον και όχι εγώ θα έπρεπε να ε, σκεφτώ να δημιουργηθεί ένα κέντρο καινοτομία, ας πούμε, που θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλαμε είναι να δημιουργήσουμε την, την Task Force, να την κάνουμε ένα είδος μόνιμης, ε, μόνιμου κέντρου ή μόνιμης εγκατάστασης, έτσι ώστε να αφιερωθούν πόροι έτσι ώστε νέοι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν έρευνα κτλ. Γι' αυτό λοιπόν... Αλλά βεβαίω θα πρέπει να υπάρξουν πόροι έτσι ώστε να συνεχίσει η προσπάθεια και να γίνει και το follow-up και η παρακολούθηση. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στην ε, υλοποίηση του, της νομοθεσίας. Νομίζω ότι ακριβώς ε, η εφαρμογή, η υλοποίηση της, ε, νομοθε, της νομοθετικής ε, νομοθεσίας, της φορολογικής νομοθεσίας είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα δυνατότητας διαλόγου και ε, ε, του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται κάποια στοιχεία από την ευρωπαϊκή δημοκρατία στην ε, εθνικού επίπεδου δημοκρατία. Και θα πρέπει βεβαίως και να πιεστεί και να οθηθεί η Κομισιόν, αλλά και από κοινοβουλευτικής πλευράς να υπάρχει αυτή η όθηση για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες. Και νομίζω ότι αν και οι δύο πλευρές ε, προωθήσουν τα θέματα αυτά, ε, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να, έχουμε, να δώσουμε στους πολίτες αυτήν την αίσθηση. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση ε, McDonald και Γενικώ, ναι, δεν ήταν επιδότηση κρατική επιδότηση, ήταν όντως μια διπλή αποφυγή φορολόγησης. Ε, και αναφερθήκατε στο πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτού του είδους τα παραθυράκια, γιατί ένα τέτοιο παραθυράκι, παραθυράκι ήταν η υπόθεση McDonald's του Λουξεμβούργου. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει διαρκώς να προσπαθούμε και διαρκώς να χρησιμοποιούμε την δημιουργικότητά μας έτσι ώστε να μπορούμε να κλείνουμε πρώτον να ανακαλύπτουμε αυτά τα κενά, αυτά τα παραθυράκια και μετά να τα κλείνουμε. Και αν ξαναεμφανίζονται να τα ξανακλείνουμε. Αυτό. Είμαστε άνθρωποι έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό ανοίγουμε διαρκώς τέτοια παραθυράκια. Δεν έχω συγκεκριμένε ιδέες για το πώς να υποστηρίξουμε την καινοτομία, την έρευνα κτλ. Αλλά οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε η Ευρώπη θα πρέπει να μείνει στην κορυφή της αξιακής αλυσίδας και να είμαστε σίγουροι ότι η τεχνολογία, η έρευνα, η καινοτομία, η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα τα παραδείγματα της ε, μικροηλεκτρονικής, ας πούμε, είναι σημαντικά. Υπάρχουν ε, ε, κοινά προγράμματα μεταξύ πέντε χωρών, Γαλλία, Γερμανία, ε, Βρετανία κλπ. Ε, και προσπαθούν ταυτόχρονα και από κοινού να προωθήσουν την έρευνα. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και μάλιστα και μια ε, προορατική ας πούμε κίνηση. Γιατί οι μεμονωμένες εταιρείες είναι λίγο δύσκολο να βρουν ακριβώς σε ποιους τομείς και με ποιο τρόπο θα πρέπει να επενδύσουν. Ε, και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κάποια καθοδήγηση όσον αφορά την καινοτομία. Πρώτα, ε, Τόμας Μάν και παρακαλώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι να μην ξεπερνάτε κατά πολύ το ένα λεπτό. Μεγάλη πρόκληση για το ένα λεπτό. Ε, κύριε Φεστάγκρεση, δικαίω σας επενούν για την ε, εργασία σας ως Επίτροπο. Το θέμα λοιπόν είναι τα φορολογικά πλεονεκτήματα για την Apple, την McDonald's και άλλα παραδείγματα που έχετε να πει. Εγώ πέρα από τις συντολογικές αυτές αρχές, οι οποίες είναι καλές στη θεωρία, αλλά δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την πράξη, έχω να ρωτήσω λοιπόν, η, η απάντησή σας σε ό,τι αφορά το Βέλγιο, για παράδειγμα. Καλέσατε το Βέλγιο να ζητήσει τα χρωστούμενα φορολογικά, τα οποία α, αναλογούν σε 700 εκατομμύρια μόνο, στο Βέλγιο. Ξέρετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Καταρχάς, οι ευρυγικές αρχές έχουν συλλέξει αυτούς τους ε, φόρους που δεν έχουν καταβληθεί στην νομοθεσία τους διευκρίνησαν ότι οι φόροι αυτοί θα μπουν σε κλειστούς λογαριασμού και θα παραμείνουν εκεί όσο του οριστικοποιηθούν οι υποθέσεις αυτές και η οριστικοποίηση δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η δικαστική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Εδώ φυσικά ε, είναι δική μου η εκτίμηση αυτή γιατί κοιτάμε ποιο θα είναι το follow-up γιατί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου περιέχει κάποια στοιχεία. Καταρχάς ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχει ακύρωση, αλλά Για κάθε πολυεθνική που προστίθεται στο σύστημα αυτό, οι βελγικές αρχές θα εκδώσουν δικαστική απόφαση για την κάθε εταιρεία. Άρα υπάρχει αυτή η ιδιωτική φύση της βελγικής αυτής, ε, του βελγικού αυτού συστήματος. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα για κάθε πολυεθνική και πάνω απ' όλα έχουμε και δικαστική απόφαση. Μετά θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Υπάρχει όμως και μια θετική πλευρά. Καταρχάς, ότι μας είπαν ότι μπορούμε να το εξετάσουμε το θέμα αυτό και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι όντω μπορούμε να το ερευνήσουμε αυτό ως θέμα κρατικής ενίσχυσης. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Κατά δεύτερον, δεν ε, ακούσαμε τίποτα για το κατά πόσο πρόκειται για κρατική ενίσχυση ή όχι. Αυτό δεν ήταν τμήμα των φιλοδοξιών τους. Και για μας λοιπόν είναι σημαντικό να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε ε, την δικαστική απόφαση και μετά να αντιδράσουμε, γιατί θεωρώ ότι έχει αποχρώσεις η δικαστική απόφαση και περιέχει πολλά και διαφορετικά μηνύματα. Αυτά θα κληθούμε λοιπόν να αναλύσουμε, να πάρουμε υπόψη πρώτα αποφασίσουμε ποια θα είναι τα μελλοντικά μας βήματα. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, η Περβάνος Euh, Ευχαριστούμε, Επιτροπέ. Με συγχωρείτε που δεν άκουσα την ε, εισήγησή σας. Ξέρω ότι αναφερθήκατε στην απόφαση του δικαστηρίου, την πιο πρόσφατη, τα είπατε, αλλά ήθελα να επανέλθω, γιατί είναι μέρος των αποφάσεων που έχουμε ανάγκη να τις δούμε και να τις ξαναδούμε για να μάθουμε απ' έξω τις λεπτομέρειες το δικαστήριο θεωρεί ότι το, σύστημα, το βελγικό σύστημα δεν είναι παράνομη κρατική βοήθεια, όμως αυτή η αρχή επέτρεψε σε κάποιες εταιρείε που είναι μέρος πολυεθνικών να αποφεύγουν φόρους στο Βέλγιο. Μετά από προηγού, πρώτερες μάλλον, ε, φορολογικές συμφωνίες και με μεγάλο κέρδος. Έτσι, έχει πληγεί η φορολογική βάση και το 2006 μόνο 30, μόνο 30 εταιρείε έκαναν χρήση φορολογικών συμφωνιών. Ε, κατηγορήθηκαν για παράνομες συμφωνίες οι Βέλγοι και επειδή αυτή η απόφαση τους αφορούσε, οι Βέλγοι θα πρέπει να παρνηθούν 242 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το γνωρίζουν πια όλοι στο Βέλγιο. δεν θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα προηγούμενο και για άλλα φορολογικά καθεστώτα με προτιμησιακέ ε, διευθετήσει. Στην περίπτωση τη Apple, λόγω χάρη. Η φορολογική δικαιοσύνη αρχίζει να αναγνωρίζεται ω πολιτικό ε, πρωταρχικό σκοπό. Τι εργαλεία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπεύεται να ασκήσετε έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου. Uh, Μπορώ σύντομα να επιβεβαιώσω ότι πρέπει κανείς να διαβάσει ολόκληρη την απόφαση και τις λεπτομέρειές της. Διότι δεν είναι απλώς αρνητική. Πρέπει να διαβάσει κανείς όλα τα τμήματα, γιατί πρώτον το δικαστήριο δεν εξέφρασε θέση ως προς το κατά πόσον οι, εται, οι αποφάσεις, οι συμφωνίες αναεταιρεία ήταν κρατική βοήθεια. Αυτό έχει παραμείνει ανοιχτό. Δεύτερον, το δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ενώ η φορολογία ε, αυτή καθεαυτή είναι θέμα των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ελέγχει τι φορολογικέ διαθετήσει για να δει αν υπάρχουν παράνομε κρατικέ βοήθειε. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Διότι οι Βέλγοι είπαν ότι αυτό δεν έχετε δικαίωμα καν να τα κουμπίσετε. Και το δικαστήριο λέει έχουμε. Έχουμε Απλώ δεν ε, τοποθετούμαστε για το κατά πόσο είναι κρατική βοήθεια ή όχι. Αυτό που είπε το δικαστήριο είναι ότι εσεί θεωρείτε ότι είναι ένα σύστημα, μια διευθέτηση. Γιατί ήταν μόνο για πολυεθνικέ. Αλλά επιπλέον για κάθε πολυεθνική που συμμετέχει σε αυτό το σύστημα, οι βελγικές φορολογικές αρχές έχουν μια ξεχωριστή φορολογική συμφωνία. Είναι δηλαδή αμφίδρομη η διαδικασία. Πρέπει κανείς να πάρει μέρος σε αυτο το συστημα οι βελγικες φορολογικέ αρχέ εχουν μια σύστημα, κανεί να παρει μέρο σε ενα συστημα αλλα και πάλι ε, ελέγχουν την κατάσταση οι φορολογικές αρχέ. Αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Διότι νομίζω ότι αυτό που ήταν ε, ξεκάθαρο και το πιστεύω ακόμα είναι ότι οι εξαιρέσεις επέτρεψαν σε κάποιες από τις πολυεθνικές να μειώσουν το φορολογήσιμο κέρδος τους ως προς 90, ως, μάλλον κατά 90%. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που είχαμε να κάνουμε με ολόκληρο σύστημα. Έχουμε ακόμα κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν κριθεί, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, που θεωρούμε ότι και αυτό είναι ένα σύστημα για συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά δεν έχει μεμονωμένες φορολογικές συμφωνίες στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι υπάρχει αναεταιρεία φορολογική συμφωνία. Και αυτό αλλάζει. Η φορολογική συμφωνία είναι για εσά, για τη δική σα εταιρεία, για τη γειτονική σα εταιρεία εκεί ή εκεί έχει άλλη συμφωνία. Είναι για εσά και μόνον. Υπό αυτήν λοιπόν την έννοια, η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ συγκεκριμένη ε, και αφορά ειδικά το πρόγραμμα του επιπλέον κέρδου. Ευχαριστούμε για του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, η κυρία ε, Ρουχόνεν Λέρνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που συμμετέχετε σε αυτήν την ακρόαση και γνωρίζουμε ότι οι κανόνες του Facebook και γενικώ της αγοράς κοινωνικών δικτύων στην Ευρώπη όλες αυτές οι εφαρμογές, τα apps που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές το Instagram, το Spotify, το Messenger, όλα αυτά έχουν σχέση με το Facebook. Βλέπουμε να ξεσπάει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και όμως αυτή η εταιρεία έχει κέρδη ρεκόρ και ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξεφύγει από το Facebook. Το Facebook ε, βασίζεται στο ότι πολλοί αισθάνονται ότι αν εγκαταλείψουν το Facebook διαπράττουν κοινωνική αυτοκτονία. Είναι πολύ δυνατοί λοιπόν και δεν έχουν και τίποτα χρήστε με ιδιαίτερα προβεβλημένου. Είναι καθημερινοί άνθρωποι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείτε ότι τα ευρωπαϊκά κοινωνικά δίκτυα, η αγορά του δηλαδή, ε, διέπεται από ανταγωνισμό υγιή ή η δεσπόζουσα θέση του Facebook είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είχαμε ακόμα υπόθεση ε, Facebook για κακή χρήση δεσπόζουσας θέσης. Ε, το είδαμε στη Γερμανία όμως ότι ε, προσπαθούν να βρουν ε, αυτό τον χώρο, αν θέλετε, όπου τέμνεται ε, η δημόσια ζωή και η ιδιωτικότητα και ο ανταγωνισμός. Επίσης το θέμα είναι ότι θα πρέπει νομικός να αποδείξεις αυτό που γνωρίζεις διαστητικά, δηλαδή ότι το Facebook ε, έχει δυσπόζουσα θέση. Και επομένως, ε, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι είναι αποδεκτό γενικά ότι το Facebook έχει δεσπόζουσα θέση, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει και νομικός να αποδεχτεί. Να Uh, uh, ναι, βεβαίως προβληματιζόμαστε και εμείς. Και ένα θέμα είναι το ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη υπόθεση ε, και άλλο είναι να πούμε ότι δεν θα έχουμε ποτέ υπόθεση Facebook γιατί εμείς παρακολουθούμε την αγορά, βλέπουμε, προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία ε, και διαφημίσεις κτλ. Και, τα λοιπά, και αυτά όλα τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Και βεβαίως και για, και άλλους παρακολουθούμε ακριβώς για τους ίδιους λόγους, ε, γιατί είναι μεγάλες εταιρείες, γιατί είναι ε, πλατφόρμες ε, και κυρίως χρησιμοποιούνται και οι πλατφόρμες αυτές και για, δημοσι... και για διαφημίσεις και επομένως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η αγορά και φυσικά η επιτήρηση γίνεται και γίνεται συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ από την Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Τόρβαλτς. Και ευχαριστώ την Επίτροπο που είναι εδώ. Στην Επιτροπή για τα Panama Papers είχαμε τον Jean-Claude ο οποίος προσπάθησε νομίζω να μας εξηγήσει ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε γιατί αυτές οι δουλειές είναι μακρόπνοες. Και κερδίζει αυτός που αντέχει περισσότερο. Αλλά βεβαίως τίποτα δεν είναι και δεν θα είναι εύκολο και αυτά που είπατε ότι ολόκληρη, στο σύνολό της δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πιέζει διαρκώς, ε, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και μακάρι να μπορέσετε να το κάνετε και να μας δώσετε και κάποια καλά παραδείγματα, περισσότερα καλά παραδείγματα. Όταν είδα την απόφαση του δικαστηρίου, αμέσως πήγα στο Google για να δω εάν κάποιος και ποιος αντιδρά και αντέδρασαν όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες στην ουσία δημιουργούσαν αυτά τα παραθυράκια για να τα εκμεταλλευτούν στο μέλλον. Θα πρέπει τώρα να δούμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι ώστε για να είναι πάντα δύο-τρία βήματα μπροστά από εσά. Γιατί στην ουσία το παιχνίδι που παίζετε κι εσείς εδώ είναι ότι προσπαθείτε να πιάσετε αυτούς που βρίσκονται ήδη δύο-τρία βήματα πιο μπροστά από εσά. Και βέβαια Όσο περισσότερα χρήματα ξεφεύγουν από τον κρατικό κορβανά, τόσο περισσότερο και οι Υπουργοί Οικονομικών και οι άλλοι Υπουργοί θα προσπαθούν και σε εθνικό επίπεδο να ε, ε, ζητήσουν βοήθεια και από τις Βρυξέλλες έτσι ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Πού βρισκόσαστε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, ε, κλέφτες και αστυνόμοι? Απάντηση. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω και με ευκολία. Ο Πιέρ Μοσκοβιτσί ήταν σεφ για το θέμα, επικεφαλής δηλαδή υπεύθυνο για το θέμα της ε, νομοθεσίας ε, ε, και βρήκε ότι τα ποσά των μη καταβληθέντων εταιρικών φόρων ήταν πάρα πολύ ψηλά. Ένας από τους λόγους που βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ έγκαιρη αυτή ε, η συνάντηση είναι γιατί βρισκόμαστε ε, στη διάρκεια της προεκλογικής στην ουσία εκστρατείας για το επόμενο κοινοβούλιο. Πρόκειται για ε, εκλογική διαδικασία στην οποία 46% του κόσμου συμμετέχει συνήθως. Άρα είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να κάνετε υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά να έχετε να δείξετε και κάποιες υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει καλά και οι οποίες έχουν λυθεί ε, ε, είτε με ομοφωνία πούμε στο Συμβούλιο. Και νομίζω ότι η πίεση που ασκείται και από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Είναι λίγο σαν να γίνεται έκκληση από, από πλευρά σας και από όλους μας ε, στους ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε ε, εδώ κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά και πρέπει και εσείς να, να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί εάν δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από πλευρά των ψηφοφόρων, τότε ούτε και εμείς θα πιέζαμε ίσως, δεν θα είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία πίεσης. Ε, γιατί όταν ε, οι πολιτικοί κάνουν καλά τη δουλειά τους, ενδιαφέρονται και οι πολίτες. Ε, στην Δανέζικη, στο δανέζικο τύπο, ε, διαβάσαμε ότι υπάρχουν πολλά συνταξιδιωτικά ταμεία τα οποία ε, πρώτα ε, προσλαμβάνουν screening experts πριν αποφασίσουν πού θα επενδύσουν. Τα κριτήρια τους είναι πολύ συγκεκριμένα και πραγματικά χτενίζουν όλη την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι πολλοί οι πολίτες που είναι αποφασισμένοι. Και το ίδιο ε, γίνεται και με την συμβολή στην κοινωνία και τον τρόπο του επιχειρήν. Και χαίρομαι γιατί συζητούμε όλα τα θέματα αυτά και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσουν και ε, περιεχόμενο της συζήτησης αλλά και περιεχόμενο της μελλοντικής εντολής. Ευχαριστώ. Thank ε, Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και καλώς ορίσατε, Επιτροπέ. Θα γνωρίζετε ότι η ομάδα μας GUNGL δημοσίευσε πέρσι μία έκθεση, μία εξέταση Τη ε, δομής της Apple μετά το 2015 σε ό,τι αφορά την έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις και φαίνεται σύμφωνα με την έρευνα αυτή ότι με την υποστήριξη της Ιρλανδικής κυβέρνησης η Apple δημιούργησε μια νέα δομή που και πάλι α, της δίνει απαλλαγή από όλα τα κέρδη εκτός, Ευρωπαϊκής, εκτός ε, Ηνωμένων Πολιτών και αυτό προφανώς της δίνει ε, μια τεράστια προβάδισμα. Ο πρόεδρος ε, του σχετικού δημοσιονομικού συμβουλίου στην Ιρλανδία επεσήμανε ότι αυτή η δομή ενδεχομένως να είναι παράνομη γιατί ο νόμος απαγορεύει τη χρήση των δομών για την φοροποφυγή και με την ίδια λογική χρησιμοποιήθηκε και τελικά για την απαλλαγή από την Ιρλανδική αμα, φορολόγηση. 2,5 ευρώ από το 2015 και μετά. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να προασπίσετε την δικαστική απόφαση σε σχέση με το πώς είχε η κατάσταση πριν το 2014 σε ό,τι αφορά και την ελληνική κατάσταση. Αλλά η πρώτη ερώτηση είναι, έχετε κάποιο χρονικό περιθώριο, κάποιο χρονικό πλαίσιο για το πότε θα λάβει η χώρα αυτή τη διαδικασία. Και κατά δεύτερον, σκοπεύετε να εξετάσετε τις νέες δομές που συστήθηκαν από πλευρά της Apple τα τελευταία χρόνια για να αποφαθείτε κατά πόσον πρόκειται για παράνομη νομική ε, κρατική ενίσχυση από την ε, Ατλαντική κυβέρνηση. Για την πρώτη ερώτηση, απάντηση. Δεν ξέρουμε πότε θα αποφασίσει το δικαστήριο για την φορολογική υπόθεση της Apple. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου που το γνωρίζουμε θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι οι Ιρλανδικές αρχές ε, ε, οριστικοποίησαν την ανάκτηση των ε, φορολογικών αυτών εσόδων τον περασμένο Απρίλιο λόγω και του ύψους των φόρων. Η νέα λοιπόν αυτή η δομή. Τι έχουμε μάθει για αυτήν. Η χρήση τέτοιων τον Capital Allowance που είναι ανοιχτό για όλες τις εταιρείε. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει σε επίπεδο κράτους δεν μπορούν να πληρώνονται οι όροι γιατί αν ισχύει αυτό για όλους απλά δεν είναι επιλεκτικό σύστημα. Άρα στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συζητήσουμε για το κατά πόσο καταβάλλονται σωστοί φόροι ή όχι. Απλά αυτό καταδεικνύει ότι σωστά γίνεται μια έρευνα για κρατικές, παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Επίτροπε. Καταρχά. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για τα όσα κάνετε τα τελευταία χρόνια. Βοηθήσατε την αποστολή τη επιτροπή μας ε, σαφώς σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή σας και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ακόμα λυπάμαι που δεν είστε η κορυφαία υποψήφια για την ομάδα της Άλντε και είναι κρίμα το γεγονός ότι δεν το έθεσε αυτό ως προτεραιότητα η Άλντε, γιατί θα ήταν φανταστικό να ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης η φορολόγηση από πλευράς της Άλντε. Πέραν τούτου όμως, θα ήθελα να κάνω και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα επόμενα βήματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Πρώτον, λοιπόν, η έκθεση Ραϊμόν σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, η ετήσια έκθεση, καλωσορίζει το γεγονό ότι η ομάδα για τι κρατικέ ενισχύσει σε ό,τι αφορά τα φορολογικά προτερήματα έχει καταστεί μόνιμο όργανο. Αυτό είναι σωστό. Αλλά και το ότι έχει τις σωστές, σωστούς πόρους για την έρευνα. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν τι είδου αναβαθμίσει μπορείτε να πετύχετε στον τομέα αυτό. Κατά δεύτερον, όταν ξεκινήσαμε με τα επιλεκτικά αυτά συστήματα, έγινε μια συζήτηση. Μια συζήτηση για το τι συμβαίνει με όλε τι υπόλοιπε εταιρείε που χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα. Μπορείτε λοιπόν να ανακοινώσετε ότι δεν θα υπάρξουν περιπτώσει μετά από τι εμπειρίε των τρεχουσών υποθέσεων, γιατί ξέρουμε ότι υπήρξαν χιλιάδες δικαστικέ αποφάσεις με στοιχεία τέτοια επιλεκτικά. Έγινε και η συζήτηση για το κατά πόσον θα υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ για δημοσιονομικέ κρατικέ ενισχύσει. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό επιτέλου να υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ για να α, μπουν σε ένα πλαίσιο κανόνων ε, αυτά που αποφασίσατε. Θα υλοποιηθεί λοιπόν αυτό επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχάς ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί. Το τονίζω. Ελπίζω ότι η φορολογία θα αποτελέσει ένα μεγάλο τμήμα του κοινοβουλευτικού διαλόγου, γιατί είναι ένα θέμα προφανές, ένα θέμα το οποίο θεωρώ είναι τόσο σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη να αποτελεί μια ήπειρο ευημερίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αν παραμείνουμε μόνο στην εταιρική φορολόγηση. Θέλουμε έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές, κυβερνήσει χωρί διαφθορά. Όλα αυτά χρειάζονται για ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον. Για την ερώτησή σα τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει σωστή εκχώρηση πόρων για την μονάδα που ασχολείται με τα φορολογικά μα ζητήματα. Αλλά προσπαθούμε να διαμορφώσουμε όλα αυτά με ευέλικτο τρόπο. Αν χρειαζόμαστε πιο πολύ κόσμο, να μπορούμε να προσλάβουμε να πιο πολύ κόσμο. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει χρειάζεται συλλογή, για παράδειγμα, στοιχείων, τεκμηρίων, προτού πετύχουμε κάτι. Μπορούν λοιπόν να δράσουν σε άλλο επίπεδο. Και χρειαζόμαστε του ανθρώπου αυτού λοιπόν που θα συλλέγουν τα στοιχεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευέλικτη μορφή εργασία για να μπορέσουμε να προωθούμε με γρήγορο τρόπο τις υποθέσει μα. Δεύτερη ερώτηση, τι γίνεται με του υπόλοιπου, Αν κοιτάξουμε το παράδειγμα των ε, LuxLeaks, Όλε αυτέ οι δικαστικέ αποφάσει τι οποίε και εξετάσαμε, δεν θυμάμαι ακριβώ τον αριθμό, 600 και κάτι, νομίζω ότι δύο τρίτα των δικαστικών αυτών αποφάσεων είχαν να κάνουν με εταιρείε χρηματοδότηση, όπου σε μία εταιρεία υπάρχει, σε έναν όμιλο υπάρχει μία εταιρεία χρηματοδότηση για να δανείζει λεφτά σε ένα άλλο τμήμα του ομίλου και να υπάρχει διανομή των πόρων αυτών σε τρίτο τμήμα του ομίλου. Εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν συμβεί αυτό, να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός αυτός για τη μετακίνηση κερδών από εκεί που δημιουργήθηκε και θα έπρεπε να φορολογείται κάπου αλλού, όπου η φορολόγηση είναι χαμηλή και ανύπαρκτη. Και εδώ είχαμε την υπόθεση της Fiat που θεωρήσαμε ότι ήταν αρκετά προφανής και ξεκάθαρη. Πέραν από την υπόθεση αυτή, μετά την υπόθεση αυτή, στο Λουξεμβούργο λοιπόν τραποποιήθηκε το σύστημα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επανάληψη τη υπόθεση Fiat. Και όλε οι δικαστικέ αποφάσει ε, που σχετίζονταν με το θέμα αυτό κατέστησαν ε, ε, ακύρε από 1η Ιανουαρίου του 2017. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν μπορεί να επαναληφθεί τέτοια υπόθεση στο Λουξεμβούργο και σε άλλο ένα κρατό μέλο που υπήρχε παρόμοιο σύστημα με το σύστημα του Λουξεμβούργου το οποίο οδήγησε στην υπόθεση Fiat και εκεί λοιπόν τροποποιήθηκε η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρουσιαστεί εκ νέου μια τέτοια υπόθεση στο μέλλον. Εμεί δεν μπορούμε και ούτε πρέπει νομίζω να κοιτάξουμε σε αυτές τις περιπτώσεις της λιτών λάξλεξ Δεν θέλετε να ανακτήσετε τους φόρους αυτούς για τις άλλες υποθέσεις, γιατί ουσιαστικά έτσι θα παραμείνουν άνηση οι όροι ανταγωνισμού. Απάντηση. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι προφανώς και εδώ ενέχεται ένα παράδοξο. Το γεγονός όμως ότι δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε και να κοιτάξουμε τις πιο προφανείς υποθέσεις. Γιατί αυτές οι προφανείς υποθέσεις, αν θέλετε, αποτελούν το καταλήτη για την αλλαγή, προκειμένου να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Αυτό σε καμία περίπτωση δε, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν οι φορολογικές ε, υπηρεσίες να επιστρέψουν ε, στις υποθέσεις αυτές για να τις εξετάσουν. Αν δηλαδή ο κόσμο ε, θεωρήσει ότι μια και ακυρώθηκε η δικαστική απόφαση μπορεί και χρειάζεται επιπλέον δικαστική απόφαση, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Για το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών τώρα, ελπίζουμε ότι στι αποφάσει για τι κρατικέ ανισχύσει δώσαμε κάποιε κατευθυντηρίε γραμμέ. Ελπίζουμε να δημοσιεύτηκαν και οι αποφάσει μα να δημοσιευτούν. Γιατί εκεί διαγράφονται σαφώς οι ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά την αρχή της κρατικής ενίσχυσης. Εξηγήσαμε ποιο, ποια είναι η στάση μας και η θέση μας και προφανώς όταν θα εκδοθεί και η δικαστική απόφαση θα προκύψουν και εκεί οι κατευθυντήριες γραμμές και ελπίζουμε τελικά όλα αυτά να συμπτυχθούν και να συναποτελέσουν ένα καινούριο πλαίσιο. Αλλά έχουμε λοιπόν και το Γενικό Δικαστήριο και στην παρούσα φάση εξετάζουμε κατά πόσο θα πρέπει να μείνουμε στην στο επίπεδο αυτό ή να, να επιβληθεί έφεση. Ελπίζω Η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε για συγκεκριμένους σκοπούς και για συγκεκριμένους λόγους. Ελπίζω ότι αυτό που θα συγκρατήσουμε όμως να είναι ότι ναι, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τέτοιε περιπτώσει παρόλο που η φορολογία αποτελεί ε, δικαίωμα των ε, κρατών μελών. Ευχαριστώ. Έχουμε και μία, ένα έτοιμο για η Είπατε, Επίτροπε, κάτι για τη Μαδέρα. Υπάρχει έρευνα που θα τη σχολιάσω μετά. Όμως στη χώρα μου, την Πορτογαλία, δεν έχουμε πάρει πίσω ούτε δεκαράκι για όλα αυτά τα φορολογικά σκάνδαλα που συζητήσαν Τώρα δεν θα μιλήσω για την ε, Μαδέρα, το Wikileaks, το Panama Papers, το Bahama, το Paradise, ούτε δεκαράκι. Για να μην πω για την ασυλία του 2012, ένα πραγματικό σύστημα για την ομοιμοποίηση της λεύκανσης του ξεπλήματο βαμικού χρήματο και το blackout, το φορολογικό blackout μεταξύ του 11 και του 15. Ε, από την Τρόικα εγκεκριμένο. Η Επιτροπή έχει συγκεκριμένε ευθύνε εδώ. Εσεί πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σα, ζητήσατε, καταρτήσατε κατάλογο με κρατημέλη που λένε τι πήραν πίσω για να δούμε κι εμεί τι κάποιοι ότι δεν έχουν πάρει πίσω ούτε δεκάρα. Ελπίζω ότι κατάλαβα. Αλλά στην περίπτωσή μας οι μη καταβεβλημένοι φόροι έχουν ανακτηθεί. Δεν είναι στους κατοικούς προπολογισμούς, είναι σε κλειστούς λογαριασμούς και έχουν καλυφθεί όλες τις περιπτώσεις. Όμως οι μη καταβεβλημένοι φόροι έχουν <laughs> ανακτηθεί. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Μήπως να το ξαναλέγατε για να καταλάβω η Πορτογαλία δεν έχει πάρει πίσω ούτε δεκάρα από τα σκάνδαλα, από τις φορολογικές αρχές. Οι άλλες κυβερνήσεις πάνε και ανακτούν ποσά. Οι Πορτογάλοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Είδαμε η Ελβετία να πληρώνει τεράστια ποσά ως αποζημίωση στην ε, ε, ε, Ισπανία, γιατί οι αρχές δουλεύουν, αλλά όχι στην Πορτογαλία. Τι έγινε με τη φορολογική αμνηστία του 2012 και με το φορολογικό blackout το ονομαζόμενο. Έγινε αποστολή και οργανώσαμε αποστολή στην Πορτογαλία γι' αυτό. Πάνω από δέκα δις απεστάλησαν στον Παναμά και στην Ουρουγουάη και αλλού. Όταν, όταν η, τράπεζα Σπίρτου Σάντου είχε ήδη καταρρεύσει και πτωχεύσει. Τι, τι περιμένετε. Δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι που θα το ψάχναμε εμείς. Διότι για τις εθνικές φορολογικές αρχές δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δουλειά τους στη θέση τους. Για μένα αυτό που με απογοητεύει ως Δανέζα είναι ότι είχαμε ένα τεράστιο σκάνδαλο όπου οι φορολογικές αρχές κατεκλάπησαν δεκάδες δις και αυτό πρέπει να το επιλύσουν στη Δανία οι δανέζικέ αρχέ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει οι Πορτογαλικέ αρχέ, όταν μιλάμε για φόρμα του εισοδήματο, οι πράγματα που δεν ήταν κρατική βοήθεια, πρέπει να ζητήσουν πίσω τα λεφτά του. Καταλαβαίνω το πάθο σα και είμαι βεβαία ότι θα είναι μέρος της προεκλογικής εκστρατεία και του πολιτικού σας αγώνα αυτό, αλλά πρέπει να το εξετάσουν οι εθνικές αρχές σας. Πολύ σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για αυτό το διάλογο που είχαμε και για τις τόσο εντελεχείς σας απαντήσεις και νομίζω ότι μπορώ να πω εκ μέρους όλους μας της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη δουλειά που έχετε κάνει και που κάνετε ακόμα για τον νόμιμο και θεμητό ανταγωνισμό. Καμιά φορά τον θεωρούμε ως κατευτονόητο. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια μόνιμη μάχη και πρέπει να ε, λειτουργεί το σύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει το χαρτοφυλάκιό σας ε, να πούμε ότι το έχετε χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε τόσο εργατικοί. Sorry, we will continue in uh, one minute. Θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε. Έχουμε λίγο μείνει πίσω στο χρόνο μας. Να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την κυρία Ινές Μαρία Μπαρντών Ραφαέλε, Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κυρίως θα συζητήσει μαζί μας με, για την πρωτοβουλία, για την ε, διπλή, για την ψηφιακή ε, ε, φορολογία που έχει υποβάλει η Ισπανική κυβέρνηση. Βέβαια, ίσως δεν προχωρήσει λόγω των πρόορων εκλογών που προκήρυξε ο Πρωθυπουργός για τον Απρίλιο. Θα το δούμε. Και βεβαίως θα μας μιλήσει και για, γενικότερα για το θέμα της ψηφιακής φορολόγησης στο σύνολό της και για όλη την Ευρώπη. Ε, κυρία Υπουργέ, μέχρι 10 λεπτά σας παρακαλώ να μας μιλήσετε ε, εν είδη εισαγωγής. Καλό σας απόγευμα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με προσκαλέσατε να μοιραστώ μαζί σας κάποιες απόψεις σχετικά με την θέση ε, που έχει η Ισπανική κυβέρνηση για την ε, ψηφιακή οικονομία. Πρόκειται ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, και ο τομέας αυτός είναι εξελικτικός και δυναμικός. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι έχουμε κάνει όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα ξεκινήσω βλέποντας λίγο πώς ε, εξελίχθηκε η συζήτηση για την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, ε, καθώς επίσης ε, και τα νομοθετήματα σχετικά με, τα, με τις γραμμικές υπηρεσίες. Θα σας δώσω επίσης και τη θέση μας όσον αφορά ε, την φορολόγηση της ε, ψηφιακής διαφήμισης που τώρα συζητιέται. Επίσης ε, θα αναφερθώ και σε κάποια άλλα σημεία φορολογικά τα οποία είναι σημαντικά για την επιτροπή σας. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, δηλαδή ψηφιακή φορολογία. Ε, πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση σχετικά με την προσαρμογή που θα πρέπει να έχει η οικονομία μας ε, και τα οικονομικά μας συστήματα προς την ε, ψηφιακή εξέλιξη. Τα φορολογικά συστήματα έχουν πλέον παλαιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι πεπαλαιωμένα απέναντι στις εξελίξεις της οικονομίας και επομένως θα πρέπει και στα πλαίσια του G20 και στα πλαίσια Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθηθούν λύσεις. Βέβαια είναι απαραίτητο ε, να υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο λύση γιατί έχουμε πολλές παγκοσμιοποιημένες πλέον μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα ε, και ε, που τελικά καταφέρνουν να κρύψουν ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους. Θα πρέπει επομένως να καταλάβουμε ότι πλέον και οι πολυεθνικές ε, και οι νέες τεχνολογίες έχουν πλέον άρει τα εθνικά σύνορα. Είναι ε, επίσης πολλές ε, οι ψηφιακές ε, πλατφόρμες οι οποίες έχουν μια τέτοια εταιρική δομή που τους επιτρέπει να πληρώνουν πολύ λίγους φόρους σε σχέση με τα έσοδά τους. Αυτό βεβαίως είναι πολύ κακό σε σχέση με τις μικρότερες εταιρείες οι οποίες έχουν τη φορολογική τους έδρα εκεί που είναι και η φυσική τους έδρα θα ε, ε, πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να καλυφθεί αυτή η διαφορά ανάμεσα στη φορολόγηση της τάξης του 23% στη μία περίπτωση με τη φυσική παρουσία μέχρι στο 5%. Ε, και ε, επομένως ε, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και το άλλο ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα της, της εταιρικής έδρας της εταιρεία που μπορεί να μην είναι ίδια με την φυσική έδρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΕΚΟΦΗΝ δεν κατάφερε να προωθήσει κάποιες ικανές λύσεις λόγω της αντίστασης ορισμένων χωρών, μιας μικρής ομάδας χωρών. Στην Ισπανία θεωρούμε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομία και δεν είναι δυνατόν ε, να απομακρυνθούν ε, οι εταιρείε από έναν πολύ σημαντικό και δραστήριο τομέα ε, που είναι η καινοτομία. Ε, να απομακρυνθούν λέω οι εταιρείε. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, με δικαιοσύνη, με δικαιοσύνη και με σωστό τρόπο να διορθωθούν αυτές οι ελλείψεις. Οι ψηφιακές εταιρείε και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα πρέπει ανάλογα με, τις, με τα έσοδά τους να συμβάλλουν στο φορολογικό σύστημα και οπωσδήποτε αυτό είναι και θέμα δικαιοσύνης απέναντι στους φορολογικούς φορολογούμενους πολίτες. Η νομιμότητα των ε, φορολογικών ε, εσόδων ε, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τους πολίτες αλλά και ε, τα κοινοβούλια. Ε, αυτό ακριβώς ε, το νομιμοποιημένο φορολογικό σύστημα που οδηγεί σε ικανές, ικανά δημόσια έσοδα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει στην διατήρηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, του συστήματος κοινωνικής προστασίας που είναι απαραίτητο και το οφείλουμε στους πολίτες μας η ασφάλεια και η ε, δικαιοσύνη απέναντι στους πολίτες ε, και η ε, δικιά τους ευζοία είναι αυτή που καθορίζει και την θέση τους και απέναντι στην Ευρώπη. Γι' αυτό διαπιστώνουμε με λύπη και προβληματισμό την ολοέν, τον ελένα και μεγαλύτερο προβληματισμό και την ολοέν και μεγαλύτερη αποστροφή των πολιτών σε σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν και στην Ισπανική κυβέρνηση εμείς θελήσαμε να προωθήσουμε ένα καινοτόμο φορολογικό ε, σύστημα το οποίο ε, είναι ικανό να αντιμετωπίσει μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και που κυρίως βασίζεται στην δικαιοσύνη ε, να μειώσουμε την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή που με ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εσόδων. Γι' αυτό υποβάλαμε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο ε, ένα νομοθέτημα σχετικά με μια μεταβατική περίοδο μέχρι ότου δηλαδή ισχύσει και ε, επιβληθεί η ενωσιακή φορολογία όσον αφορά αυτήν την φορολόγηση της ψηφιακής ε, οικονομίας. Το ε, βασιζόμαστε ε, στην ε, ενδελεχή ανάλυση αυτών των τριών εκατομμυρίων χρηστών που χρησιμοποιούν την φορολογική πλατφόρμα και μέσα από ένα πιο καινοτόμο σύστημα το οποίο δίνει φορολογικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες ε, οι οποίες δίνουν την ε, δυνατότητα σε εταιρείες ε, να φορολογηθούν, αποφεύγοντας όμως την διπλή φορολόγηση, ακόμα και όταν η έδρα τους δεν βρίσκεται στην Ισπανία. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε ότι ένα δις 200.000 ευρώ θα εξοικονομηθούν και θα είναι ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου αντιστοίχων εσόδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε περίπτωση δε που η οδηγία αλλάξει, ενώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τότε θα τροποποιήσουμε και εμείς ε, την δικιά μας νομοθεσία. Ε, εμείς θέλουμε να επιτύχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συνένεση όσον αφορά τα θέμα αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είναι δυνατόν τέτοιου είδους φόροι να εκφεύγουν της ε, εθνικής μας ε, αρμοδιότητας. Στην Ισπανία θεωρούμε ότι θα πρέπει να λυθούν επιτέλους τα προβλήματα αυτά. Με αυτά τα φορολογικά έσοδα και με κάποια άλλα συνοδευτικά μέτρα η Ισπανική κυβέρνηση προτίθεται ε, να χρηματοδοτήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες ε, λόγω χρόνων λιτότητας έχουν μείνει πίσω. Η, βεβαίως ε, η πολιτική κατάσταση στην χώρα μας ανάγκασε να προκηρύξουμε εκλογές για τον Απρίλιο. Βεβαίως θα συνεχίσει και μέχρι τότε η μελέτη του θέματος, έστω και αν θα σταματήσει η συζήτηση ενώπιον του νόμου αυτού, ενώπιον της ε, ε, Βουλής ε, της Ισπανίας. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας για μείωση της φορολογίας στις ψηφιακές διαφημίσεις. Θεωρούμε ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση γιατί θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην εσωτερική αγορά λόγω έλλειψης εναρμόνισης. Υπάρχουν ήδη ε, αυτοί οι οποίοι έχουν ε, ήδη δηλώσει την ε, μη συμφωνία τους όσον αφορά το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, το ποσοστό ε, του 0%. Ε, Μηδενικό λοιπόν να είναι το ποσοστό από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην βρούμε απλώς κάποιες μεσοβέζικες λύσεις αλλά να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε σωστά. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο στη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, λύσεις οι οποίες θα είναι μακροπρόθεσμες. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ε, ότι υπάρχει και η ε, νομοθεσία σχετικά του 2017 για τον ΦΠΑ και εκεί θεωρούνται οι πλατφόρμες ως παθητικές οντότητες. Επίσης και με το πρωτοβουλία της Ισπανίας οι πλατφόρμες θα πρέπει να δίνουν όλα τα στοιχεία στις δημόσιες αρχές. Υπάρχει λοιπόν ε, ε, ε, π.χ. στην Ισπανία υποχρέωση δήλωσης των τουριστικών ενοικιάσεων. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την μεταβατική περίοδο. Ε, βεβαίως θα είμαι και στη διάθεσή σας να συζητήσετε μαζί μου και οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αναφέρθηκα προηγουμένως ε, στην ε, πρόταση της ε, Κομισιόν η οποία δεν έγινε δεκτή λόγω αντίθεσης μιας μικρής ομάδας χωρών. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η μη ύπαρξη πλειοψηφικής απόφασης και η δυνατότητα βέτο ή άσκησης αρνησικυρίας από πλευράς των κρατών συχνά οδηγούν τελικά σε τελμάτωση των συζητήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να είναι πραγματικά παγκόσμιος πρωταγωνιστής και παγκόσμιος παίκτη, ε, θα πρέπει για θέματα τουλάχιστον σημαντικά όπως είναι ας πούμε η φορολόγηση ή όπως είναι ε, ε, οι πολιετής προϋπολογισμοί να εφαρμόσει την ε, πλειοψηφική απόφαση. Βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι σε φορολογικά θέματα θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν πλειο ψηφικές αποφάσεις για θέματα όπως είναι ας πούμε ε, η καταπολέμηση του ξεπλήματος και της ε, ξεπλήματος παράνομου χρήματος καθώς επίσης ε, και της φοροδιαφυγής. Η Ισπανία επίσης συμπεριλαμβάνεται στις χώρες αυτές οι οποίες συμφωνούν με το μηχανισμό ενισχυμένης συνεργασίας. Εμείς εμπνεόμενοι και από τον αντίστοιχο μηχανισμό της Γαλλίας έχουμε πάρει αποφάσεις όσον αφορά τις εταιρείες οι οποίες είναι ε, ε, ε, γεγραμμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται δεν υπόκεινται η γνώμη οπωσδήποτε σε φορολογία που θα ξεπερνάει το 0,2% σε περίπτωση που τα έσοδά τους είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Στα πλαίσια της έμεσης επίσης φορολόγησης έχουμε ε, πάρει κάποια καινούργια βήματα, τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συντονιστούν με τα όσα αναφέρονται στην ενισχυμένη, στον ε, μηχανισμό ενισχυμένη συνεργασία. Ε, τα χρήματα από όλους αυτούς τους μηχανισμούς οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθούν για βελτίωση του κράτους ε, κοινωνική μέρημνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε τελικά ένα σύστημα σωστής και αποτελεσματικής εταιρικής φορολόγησης. Και χαιρόμαστε γιατί έχει προχωρήσει η εργασία όσον αφορά το θέμα αυτό στι επαφέ με τις Τρίτε ε, χώρες καθώς επίσης και με, συνεργασί... με χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται καλά όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Καθώς επίσης ε, και θεωρούμε ότι θα πρέπει η λεγόμενη γκρίζα ε, λίστα να επικαιροποιηθεί. Λαμβάνοντα υπόψη ε, τα τελευταία ε, στοιχεία. Επίση να σας πω ότι η Ισπανία δεν βρίσκεται στην, ε, στον κατάλογο των χωρών οι οποίε έχουν δώσει ιδιαίτερες φορολογικές, ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα, καθώς επίσης και χώρες οι οποίε έχουν προχωρήσει σε ειδικέ φορολογικές ρυθμίσει. Θεωρούμε όμω ότι ένα καλό βήμα θα θα ήταν ε, να υπάρχει ενιαίο ποσοστό εταιρική φορολογίας για ε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, κύκλο εργασιών πάνω από 20 εκατομμύρια. Οπωσδήποτε με, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρές εταιρείε, τις μικρές επιχειρήσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τον ανταγωνισμό τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά την έννοια αυτή θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και να σας πω λοιπόν ότι η Ισπανία ε, συμφωνεί ε, με την προτινόμενη τροποποίηση της 34-2013. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υποστηρίξω και να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πρέπει με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε απέναντι στις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ε, να συμβαίνουν τέτοιες ε, ε, παραβιάσεις όσον αφορά την φορολόγηση. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, ε, ενοποιηθούν οι φορολογήσεις είτε πρόκειται για το σύστημα ΦΠΑ είτε πρόκειται για, τις, ε, για, την για, τον φόρο των εταιριών. Οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και το συμφέρον του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα υπάρχουν πολλές διαφορές και λέμε ότι μονάχα θα είναι είναι δυνατή η Ευρώπη αν καταφέρει να προχωρήσει ενωμένη. Και θα προχωρήσει μονάχα η Ευρώπη εάν μπορέσει να δώσει στους ε, ε, πολίτες της ελευθερία, δικαιοσύνη ε, και επομένως δικαιότερη και πιο διάφανη και πιο προοδευτική φορολογία και αντίστοιχα φορολογικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο διεξοδική παρουσίαση της σφαιρικής αυτής προσέγγισης. Τώρα θα έχουμε τη συζήτηση με τα μέλη. Ο καθένα θα έχει πέντε λεπτά για να θέσει την ερώτησή του και να λάβει την απάντησή του ταυτόχρονα. Ένα λεπτό η ερώτηση, τέσσερα λεπτά η απάντηση. Να ξεκινήσουμε με τον συνεισηγητή μας για το ΕΛΚ, τον κύριο Νίντερμαγερ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Μια απλή ερώτηση. Γιατί δυσκολεύτηκατε τόσο να συμφωνήσετε για τα πιο σημαντικά φορολογικά ζητήματα, όπως τον ε, ψηφιακό φορό, το CCCTB και το BAT. CTB μάλλον. Και γιατί δεν προχωράτε σε μια πιο ενισχυμένη συνεργασία στα φορολογικά ζητήματα, όπως πολλοί θα περίμεναν. Bueno, respecto al acuerdo... Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, η δυσκολία δηλαδή επίτευξης ε, συμφωνίας, όπως είπα και προηγουμένως, πραγματικά είναι σοβαρή η δυσκολία εξισορρόπησης της ε, αυτονομίας ή της ευθυνικής κυριαρχίας των χωρών ε, από την μία πλευρά και την ενωσιακή ας πούμε διάσταση. Θα πρέπει να γίνονται επομένως, αμοιβέ υποχωρήσεις, αλλά ε, να λαμβάνονται και οι αποφάσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα να προωθηθούν ενιαίες λύσεις. Η συνένεση βεβαίως έρχεται μετά από χρόνια. Σε μερικές περιπτώσεις τουλάχιστον είχαμε και 8 ε, χρόνια στην ε, Ισπανία. Θεωρεί ότι πλέον ε, δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε αυτήν την απαραίτητη ψηφιακή δικαιοσύνη γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή. Αλλάζει η οικονομία, αλλάζουν οι συνθήκες, όπως είπα και προηγουμένως, δεν ε, ε, γνωρίζει όρια και σύνορα η οικονομία, δεν παίζει πλέον τόσο ρόλο και δεν είναι περιοριστική η έννοια της έδρας μιας επιχείρησης και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε με επαναστατικό, νεοτεριστικό τρόπο. Γιατί η αλλαγή των συνθήκων της οικονομίας ε, σημαίνει ότι θα πρέπει βάθρων να αλλάξει και το φορολογικό μας ε, σύστημα. Η Ισπανία είναι ένα κράτος το οποίο βεβαίως ε, θέλει και την αμοιβαία αρρωγή και τους μηχανισμούς βοήθειας. Δουλεύουμε πάντα για την μεταφορά όλων των ε, νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταφορά ε, στο εθνικό επίπεδο. Κύριο Σκόφου για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρα και ευχαριστώ και την Υπουργό που ήρθε στην Επιτροπή μας και εξήγησε την σημασία το να υπάρχει ένα σύστημα για το σοφόρο των εταιριών που να είναι προσαρμοσμένο στι ανάγκε του 21ου αιώνα και την σημερινή οικονομία. Συμφωνώ απολύτω με την Υπουργό ότι αν αυτό δεν το λύσουμε τώρα, έχουμε άμεση απειλή για το σύστημα των κρατικών βοηθών στην Ευρώπη και το κατά πόσο θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε το σύστημα κοινωνική πρόνοια. Η ερώτηση μου αφορά και πάλι τη φορολογική, την ψηφιακή μάλλον φορολογία. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε, διότι μια από τι επιφυλακτικότερε κυβερνήσει είναι η Δανέζικη. Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις τους, όμως επιχειρηματολογούν ότι φοβούνται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από την πλευρά των Αμερικανών εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εφαρμόσει εταιρικό φόρο για τα ψηφιακά. Ποια είναι η δική σας άποψη. Είμαστε δυνατοί, αρκετά δυνατοί για να έχουμε μια ενιαία θέση εδώ και σε συνεργασία με άλλες μεγάλες οικονομίες και δεύτερον, η ομάδα του κώδικα συμπεριφοράς για την ε, εταιρική φορολογία. Αυτή η ομάδα υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη πρόοδου στα φορολογικά στην Ευρώπη εδώ και χρόνια και το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή έχει πολύ άμεση επαφή με άλλες ομάδες στο Συμβούλιο και με το Διαμεσολαβητή. Ε, και ο Διαμεσολαβητής μάλλον το έχει εντοπίσει αυτό. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι και στην επίπεδο αυτή τη ομάδα για να μπορούν και τα μέσα και ο κόσμο να παρακολουθεί τι συμβαίνει και να ξέρουν ποιο μπλοκάρει τι. Γιατί για τα θέματα αυτά απαιτείται ομοφωνία. Αλλά σίγουρα μπορεί κανείς και, και κλεισμένο των θυρών να μπλοκάρει την πρόοδο κάποιες ε, χρήσιμης νομοθεσία. Sí, gracias. Bueno, Σας ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση που μου απευθύνετε Γιατί αυτό που είπατε, ε, δηλαδή... Ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον ε, φόρο αυτό. Πιστεύω ότι η συζήτηση γίνεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Ε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε ε, βράχη πρόθεσμα και τι μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα Σε αυτήν την περίπτωση όμως οι Ηνωμένε Πολιτείες βρίσκονται στην ίδια θέση ε, και προβληματίζονται και αυτές λόγω της αλλαγής της οικονομίας και για την αλλαγή της οικονομίας γιατί αυτό, αυτή η αλλαγή γίνεται παγκόσμια. Και Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα βράχη πρόθεσμα και ε, μακροπρόθεσμα. Βράχη πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Ε, η Ισπανία σε, αυτή την, ε, αυτό το θέμα συμφωνεί με πολλές άλλες χώρες και επομένως λέει ότι θα πρέπει οι στρατηγικές βραχυπρόθεσμες αντιμετώπισης θα πρέπει να συνδυάζονται και να εντάσσονται σε ένα μακροπρόθεσμο ε, πρόγραμμα και σχέδιο. Και επομένως, οπωσδήποτε, θα πρέπει η, τα έσοδα των μεγάλων αυτών εταιριών να μοιράζονται με κάποιο τρόπο και ισομερός ε, στις ε, χώρες στις οποίες έχουν παρουσία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ποια είναι τα κριτήρια αυτά ε, ε, τα οποία θα μας οδηγήσουν μέσα από κάποια ενδιάμεσα μεταβατικά μέτρα στα τελικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν και στην τελική λύση σε παγκόσμιο συνολικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε όλες τις ε, δυνατές λύσεις έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε αυτήν την τελική λύση. Στην Ισπανία ε, η συζήτηση ήταν πάρα πολύ έντονη όπως γνωρίζετε, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει η συζήτηση αυτή. Και εν τέλει είχαμε μια εκπληκτική συνένεση. Μας ε, κατέπληξε αυτή η συνένεση γιατί ε, εμείς ήρθαμε σε επαφή με πολλούς εμπλεκόμενους από την τεχνολογία, από την αγορά και τα λοιπά και πραγματικά συμφώνησαν όλοι respecto de los, de los contribuyentes. Respecto de la segunda pregunta. De... Όσον αφορά την ερώτησή σας ε, για, το, για την ομάδα δεοντολογίας, ε, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την ερώτησή σας, αλλά να σας πω ότι σε αυτήν την ε, ομάδα γίνεται δουλειά. Ε, βέβαια, ναι, είναι αλήθεια ότι η ισορροπία μερικές φορές είναι περίπλοκη έως πολύ περίπλοκη γιατί τα θέματα που τους απασχολούν είναι ευαίσθητα, τα έγγραφα εργασίας επίσης είναι πολύ ε, ευαίσθητα, γι' αυτό και, και πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια Οπωσδήποτε η Ισπανία θέλει να προωθηθεί η ε, διαφάνεια όσον αφορά αυτήν την ε, ομάδα. Υπάρχει επίσης ε, και υπάρχουν και τα επεξηγηματικά δελτία όσον αφορά τις δραστηριότητες της ομάδας αυτής. Αλλά τώρα η αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων είναι λίγο πιο δύσκολο όντως. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τα όρια τα οποία έχουν, ε, ε, τα, να γίνονται σεβαστά τα όρια τα οποία οι χώρες θέτουν ε, για λόγους σεβασμού της εθνικής τους κυριαρχίας όπως λένε. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Χωσέ Σαλαφράγκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Το Κοινοβούλιο δεν δέχτηκε τους προϋπολογισμούς. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι τα προβλήματα είναι συνολικά και ε, παγκόσμια και τέτοιες λύσεις θα πρέπει να βρούμε και θα πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ε, Ε, η Ισπανία βρίσκεται στο, ε, στο σημείο ε, 36 από 63 χώρες. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε περισσότερο τους δείκτες έτσι όπως αυτοί έχουν οριστεί από χώρες πιο προχωρημένες όπως είναι η Δανία ή η Σουηδία. Επίσης όσον αφορά τα οικονομικά κημητήρια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια συζήτηση και όσον αφορά το θέμα αυτό. Απάντηση. όσον αφορά το πρόβλημα. Ναι, τα προβλήματα είναι συνολικά, είναι παγκόσμια, άρα θέλουμε και παγκόσμιες λύσεις. Αλλά όταν η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί προβλήματα ή βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, ε, τότε θα πρέπει να ε, βρούμε κάποιες ε, κινητήριες δυνάμεις για να τραβήξουν μπροστά την κοινωνία. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Ισπανία και βέβαια δεν είναι μονάχα η Ισπανία η οποία έχει πάρει αποφάσεις όσον αφορά ας πούμε φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κλπ. En todo momento cuando se ha hecho un planteamiento de estas dos... και η Ισπανική κυβέρνηση ε, πήρε κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε πραγματικά να αποτελέσει κινητήρια δύναμη και μοχλό ε, για την ε, και μοχλό για την οικονομική πρόθεση. Και μακάρι να είχε προκύψει ε, συνένεση. Κοιτάξτε, ε, αυτή η, αυτός ο φόρος είναι μόνο 3% και οπωσδήποτε λαμβάνει ε, υπόψη το γεγονός ότι αναφέρεται σε έναν τομέα ο οποίος δεν είναι επιβαρημένος. Είναι λογικό ε, ότι εδώ υπάρχει μία καινοτομία ε, και ε, τουλάχιστον δίνει κάποια λύση ή αντιδρά σε μια κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει ήδη από καιρό γιατί δεν είναι και τόσο πρόσφατη κατάσταση. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε αυτές τις λύσεις οι οποίες μπορεί να μην έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνένεσης αλλά ε, παρόλα αυτά πρέπει να ε, προχωρήσουμε. Όσον αφορά τώρα τον ε, προϋπολογισμό, να σας πω ότι ο προϋπολογισμός της Ισπανίας είχε καθαρά κοινωνικό προσανατολισμό και τα έσοδα είναι αυτά τα οποία θα μας επέτρεπαν αυτόν τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Ε, και από την άλλη πλευρά, ε, οπωσδήποτε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τους ε, κανόνες της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αλλά να σας πω ότι αυτό που μας απασχόλησε, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες και τα έσοδα, ε, αυτό που μας απασχόλησε, λέω, είναι να έχουμε ένα προϋπολογισμό ε, ο οποίος να απευθύνεται και να λαμβάνει υπόψη τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ραμόν Χαουρέγγι. Ε, να σας ευχαριστήσω πολύ ε, για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε τη θέση της Ισπανίας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά, έστω και αν είναι πολύ ε, εύκολο να θεωρήσει κανείς ότι συμφωνείτε με αυτά που, έχουν, ε, που έχετε κάνει, παρόλα αυτά θεωρώ ειλικρινά ότι η Ισπανική κυβέρνηση ανέλαβε τρεις φορολογικές πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές που δεν τολμούν να πάρουν άλλες χώρες Πρώτον, για το θέμα της ε, φορολόγησης, της ψηφιακής φορολόγησης ε, και να σας ρωτήσω ε, τι έγινε με τους επιχειρηματίες, τι, τι έκαναν όταν τους είπε η Ισπανική κυβέρνηση ότι θέλει να διατηρήσει αυτό το ποσοστό. Αυτές οι φορολογικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, ε, νομίζω, κυρία Υπουργέ, ότι αποτελούν και μια υπόσχεση για το μέλλον. Στις επόμενες εκλογές ενδεχομένως θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι αν εσείς επανεκλεγείτε θα διατηρήσετε τις ίδιες προτάσεις. Δεύτερον, πώς λειτουργεί το ελάχιστο ποσοστό, το ελάχιστο επιτόκιο, ε, σε σχέση με αυτό ας πούμε το 9% αυτοί που πλήρωναν 9% μπορεί να, να, χρειαστεί ε, είναι πιθανό, ας πούμε, κάποιος που πλήρωνε με συντελεστή 9% ξαφνικά να κάνει ένα άλμα ε, του, της τάξης του 6% αυτός ο συντελεστής και να φτάσει να πληρώνει 15% από τη μια μέρα στην άλλη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα όσα με όσα αναφέρατε. Πρώτον, ε, πώς αντέδρασε ο επιχειρηματικό κόσμος. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία, ε, γιατί ε, αυτή η συζήτηση έγινε σε μία εβδομάδα αναταραχών. Ωστόσο, στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής ήταν σαφής η φορολογική συζήτηση και εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους. Όμως ε, η κυβέρνηση ε, ήξερε πολύ ξεκάθαρα τι θέλει και που θέλει να πάει. και ε, δεν, ήταν σαφές επίσης ότι δεν θέλει να αγγίξει την φορολογία φυσικών προσώπων, δεν ήθελε να αγγίξει τον ΦΠΑ και δεν ήθελε να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ε, κάποιο, κάποιες οντότητες. Ε, γι' αυτό... Ε, θελήσαμε να δουλέψουμε ε, περισσότερο ε, με ε, φορείς που δεν είχαν την, όπως την ψηφιακή φορολόγηση ή όπως ας πούμε την φορολόγηση των δημοσιονομικών των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, πρόκειται για στοιχεία τα οποία αφορούν μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ε, ωστόσο, ε, είχαμε μέχρι τώρα μέχρι τώρα την ε, ιδιότυπη κατάσταση ενώ να αναγνωρίζονται ε, τα έσοδα να μην υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης τμήματος των εσόδων αυτών μέσω της ε, φορολόγησης. Εμείς Προσπαθήσαμε λοιπόν να βασιστούμε και με αυτό τον τρόπο λειτουργήσαμε ε, με έναν ε, ελάχιστο ε, συντελεστή όσον αφορά την λογιστικά φορολογήσιμη βάση. Ναι, είναι γεγονός ότι ε, κάποια εταιρεία η οποία μέχρι τώρα φορολογείται με 9, 10, 11% θα φορολογηθεί με 15%. Τώρα, ποια ήταν η αντίδραση από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ε, κάποιος, κάποια φασαρία κατά κάποιο τρόπο στη διάρκεια της ε, εβδομάδας των συζητήσεων, αλλά εμείς ε, δημιουργήσαμε το φόρουμ των μεγάλων επιχειρήσεων για τις, ε, στα πλαίσια της, του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να εξηγήσουμε ακριβώς αυτή τη μεταρρύθμιση. Και εμείς το παρουσιάσαμε ακριβώς ε, σαν μια δυνατότητα, σαν μια ευκαιρία να ανακτήσει ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας ε, την χαμένη του νομιμοποίηση. Γιατί είναι γεγονός ότι έχασε την νομιμοποίησή του τα τελευταία χρόνια. Και εμείς το παρουσιάσαμε λέγοντάς τους ότι στη ζωή κάποιες δυσκολίες θα πρέπει να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Όπως είπα και στην αρχή, ε, η κυβέρνησή μας αυτό που θέλει ε, είναι να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα διατηρήσουμε αυτήν την ε, πρόταση. Βεβαίως δεν ήταν εύκολη η κατάσταση, βεβαίως δεν ε, ήταν εύκολο να βρούμε ε, συμφιλιωτικές λύσεις μεταξύ όλων των πλευρών, ωστόσο θα διατηρήσουμε αυτήν την γραμμή. Ευχαριστώ από την Γκουε Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Όταν μιλάμε στις στα ευρωπαϊκά όργανα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε ε, την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Είναι σαν να έχουμε λίγο τον ελέφαντα στο μέσο του δωματίου και να μην τον βλέπουμε. Ναι, υπάρχουν φορολογική παράδειση εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν είναι όρις ε, ε, δεν είναι έτσι ελάσσονο σημασία. Το Λουξεμβούργο, η Μάλτα είναι μεγάλη φορολογική παράδειση. Είναι και η Ανδόρα, είναι και οι άλλες γειτονικέ χώρες όπως είναι η Ελβετία ας πούμε. Επίσης πώς μπορεί να, ε, ε, να συζητηθεί το θέμα του Brexit σε σχέση με τον αντίκτυπο στους φορολογικούς παραδείσους, αλλά ε, στις στους καταλόγους που κάνει και η Κομισιόν και οι χώρες περιέργως δεν περιλαμβάνονται φορολογική παράδειση που αφορούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχους καταλόγους των ε, διεθνών οργανισμών ε, γιατί ε, εμείς μιλήσαμε για τις Μπαχάμες, για τον Παναμά, για το Μονακό και τα λοιπά, ενώ ας πούμε και η Ιντερπολ και η οργάνωση των Ισπανών λογιστών αναφέρεται στη Μάλτα, στην Ανδόρα, στο Λουξεμβούργο ως φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν ναι, εάν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να αναφέρονται. Πώς αξιολογείτε εσείς τον ε, κατάλογο ε, αυτών των ε, φορολογικών παραδείσων. Τέλος, εσείς θα προωθήσετε ε, την, ε, τα κριτήρια τα οποία λειτουργούν, τα οποία χρησιμοποιούν άλλοι διεθνείς οργανισμοί ή το συνδικάτο που ανέφερα προηγουμένως, εσείς σκέφτεστε ε, το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τα ίδια κριτήρια. Eh, Απάντηση. η Ισπανία οπωσδήποτε ε, είναι αποφασισμένη να κάνει το πάνε έτσι ώστε ε, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινή λίστα ε, με τις μη συνεργάσιμες χώρες. Και εμείς έχουμε νέο εθνικό κατάλογο των... Θα, μάλλον θα λάβουμε υπόψη τα στοιχεία αυτά στο νέο εθνικό κατάλογο ε, ε λαμβάνουμε υπόψη όλα τα στοιχεία όπως ανέφερα προηγουμένως της ε, ε αμοιβαία αρρωγής ε, και οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει όλους τους μηχανισμούς που θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής κτλ. Τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές πρόοδους ας πούμε αυτοματοποιημένη ε, ανταλλαγή πληροφοριών, πληροφορία αναχώρα κλπ. Ε, ε, και με τον τρόπο αυτό καλύπτονται πολλά από τα προβλήματα τα οποία τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδεικνύουν. Αλλά πρέπει πάντα να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Στην Ισπανία η κυβέρνησή μας όντως ε, έχει εκδώσει μια βελτιωμένη έκδοση ε, ε, των δυνατοτήτων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης. Και βεβαίως τα κριτήρια που περιλαμβάνονται εκεί είναι αυστηρά, είναι αντικειμενικά και ακριβώς αναφέρονται στον αμερόληπτο τρόπο με τον οποίο οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να δημιουργούνται. και εμείς ε, είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία όλων των διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά όταν δημιουργούμε, όταν ε, θεσπίζουμε αυτούς τους ε, καταλόγους. Επιμένω ότι εμείς θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σωστούς ε, τέτοιους καταλόγους. Εσείς ε, αναφερθήκατε και στο Brexit. Για μας εμείς δηλαδή θεωρούμε ότι είναι και μια ε, ευκαιρία συζήτησης γιατί με, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ευκαιρία να γίνουν ε, και ε, κάποιες συμφωνίες και κάποια memorandum of understanding με το Γιβραλτάρ όσον αφορά βέβαια φορολογικά ζητήματα. Presidente, Presidente, solo una cosa. Κάτι ακόμα. Δεν μου απαντήσατε όμως. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν φορολογική παράδειση εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι θέμα που μας απασχολεί στην Επιτροπή. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση, η κυβέρνηση πιστεύει ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως ε, φορολογική παράδειση το Κοινοβούλιο έχει απαντήσει θετικά στην ερώτηση αυτή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιους, κάποια αντικειμενικά κριτήρια βάσει αυτών των κριτηρίων. Εάν διαπιστώσουμε ότι μια χώρα πρέπει να μπει σε αυτόν τον κρύο κατάλογο γιατί δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα οποία αντικειμενικά έχουν θεσπιστεί, τότε ναι. Το θέμα εδώ δεν είναι να ακολουθήσουμε τη, διεύθυνσή μας ή να πούμε ότι πιστεύουμε το ένα ή το άλλο διαισθητικά. Όχι, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε κάτι τέτοιο να καταστεί δυνατόν. Efectivamente, aplicados los criterios, ese es el resultado, pues lógicamente todos los tendremos que aceptar y que respetar. Αυτά. Και υπάρχουν αρχέ οι οποίε πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ο Σβέν Γκίγκολ για του πράσινου. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Γιατί? Μετά από εξέταση 19 χρόνων συμπεριφορά σε, ε, σε ψηφοφορία. Ε, υπάρχει μια παράδοση της Ισπανίας ε, κατά της φοροαποφυγής, υποστήριξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και φοροαπάτης. Ωστόσο, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο προφανώς προκαλεί διαφλονικία. Αυτός ο μαύρος, αυτή η μαύρη λίστα για την, το ξέπλυμα χρήματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν υπέβαλε τη δική της αξιολόγηση και τα κριτήρια τα δικά της και με μια πιο αυστηρή λίστα πλέον. Και ακούω επανελειμμένα ότι η δική σας κυβέρνηση κάνει λόμπινγκ για να βγει ο Παναμάς από τη λίστα αυτή, παρά το γεγονός ότι εδώ υπάρχει γερό προηγούμενο, γιατί ο κ. Πατέρα πριν από κάποια χρόνια έβγαλε τον Παναμά από τη λίστα των φορολογικών παραδείσεων και τώρα η, η Ισπανική κυβέρνηση ζητά από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει τον Παναμά από τη λίστα για τις χώρες για ξέπλυμα χρήματος. Και η κυβέρνηση ίσως αναζητά ειδική πλειοψηφία για να μπλοκάρει την πράξη κατεξουσιοδότηση για τη νέα λίστα. Ερωτώ λοιπόν, μπορείτε να δεσμευτείτε σήμερα να επιβεβαιώσετε σήμερα ότι δεν θα δημιουργήσετε μια πλειοψηφία κατά μια τέτοια λίστα με χώρε ξεπλήματο χρήματο. Δεσμεύεστε ότι στο μέλλον θα προσπαθήσετε να γίνετε καλύτεροι αντί να προσπαθείτε να φτιάξετε πλειοψηφία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και άλλε χώρε για να μην καταρτιστεί μια τέτοια λίστα. Bueno, ότι το είπα ξεκάθαρα προηγουμένως. Απριόρι ε, δεν υπάρχει κάποια θέση όσον αφορά το θέμα του Παναμά και για το ξέπλυμα αλλά και για οτιδήποτε άλλο Υπάρχ, πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μια χώρα μπαίνει ή όχι από, από τον κατάλογο. Όταν λοιπόν θα έχουν καθοριστεί, θεσπιστεί τα κριτήρια αυτά, τότε θα είμαστε αυστηροί όσον αφορά ε, τον σεβασμό και την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Και όταν ξεκινήσαμε το προσχέδιο νόμου, γνωρίζαμε τα στοιχεία αυτά και ακριβώς είπαμε ότι ε, ε, στον Εθνικό Κατάλογο Εθνικών στην στον Εθνικό Κατάλογο Φορολογικών Παραδείσων, ε, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Όταν θα γίνει λοιπόν ε, η επικαιροποίηση των ε, καταλόγων εδώ, θα μεταφερθούν και στους εθνικούς καταλόγους. Κατά την άποψή μας, ο Παναμά τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για ευθυγράμμιση με τις ε, αρχές και τα κριτήρια. Βέβαια, θα συζητηθεί το θέμα αυτό στην ε, Επιτροπή και οπωσδήποτε όταν ε, ε, έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οπωσδήποτε η Ισπανία θα το λάβει υπόψη και οπωσδήποτε, ε, άσχετα από ποια χώρα, για ποια χώρα πρόκειται, θα εφαρμόσει τα όσα αναφέρονται. Πρόεδρε, ο κ. η ερώτησή μου ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Θα υποστηρίξετε η λίστα αυτή να μην περάσει ως έχει τώρα ή προσπαθείτε στην παρούσα φάση να βρείτε μια πλειοψηφία που να μπλοκάρει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Ρωτώ κατά πόσον η κυβέρνησή σας θα επιτρέψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσει, κατά πόσο προσπαθείτε να μπλοκάρετε αυτή την λίστα κατά του ξεπλήματος χρήματος όσο έχει τώρα. Μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον, αλλά αυτή τη λίστα θα την μπλοκάρετε ή θα την αφήσετε να περάσει. Όχι, από όσο γνωρίζω δεν προσπαθούμε να μπλοκάρουμε καμία απόφαση τέτοια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. Ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις αποφάσεις και τις ε, διεργασίες των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση. Ο προέδρο ευγενικά Ευχαριστώ και τους διερμηνείς.